Επαναλαμβάνεται η διακοπή σε συνεδρίαση. Τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι από ό,τι φαίνεται. Ούτως λοιπόν εγκρίνονται και ακολουθούν οι σημασία σημασιας σημασίας επερωτήσεις, άρθρο 130β του κανονισμού,